Uh, Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Η συζήτησή μας είχε να κάνει με το χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα Πλαίσιο 9, πολύ σημαντικό για όλους εμάς, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και φυσικά θα ξεκινήσουμε και τη συζήτηση στην Επιτροπή μας. Να καλωσορίσω ένθερμα τον κύριο Κάρλος Μέντος, τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Έρευνα, Επιστήμη και την Κοινοτομία. Και συζητούμε σε συνεδρίαση Ήτρε όλα τα θέματα στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου φυσικά. Πιο συγκεκριμένα θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερο για την ε, ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε σχέση με την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση του ορίζοντα 2020. Επιπρόσθετα, η πρόταση για το πρόγραμμα πλαίσιο 9 θα δημοσιευτεί στα τέλη Μαΐου, ελπίζουμε. Ίσως ε, και δύο εβδομάδες νωρίτερα θα ήταν σημαντικό, το πρώτο ημίση του Μαΐου δηλαδή και τι θα μείνει το ίδιο σε σύγκριση με τον οριζόντα 2020 και τι θα βελτιωθεί. Δηλαδή, ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ τη γενική πρόταση του Ορίζοντα 2020 και τη νέα πρόταση για το πρόγραμμα Πλαίσιο 9. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να προετοιμαστούμε για τα ζητήματα αυτά και φυσικά να δούμε και την αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020. Πρόγραμμα εργασία 2018 μέχρι το 2020, του Ορίζοντα 2020, για να ακούσουμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εφαρμόζει τις προτεραιότητες της βασικής πράξης, είναι εντός του χρονοδιαγράμματος ε, αυτή η εφαρμογή και θα θέλαμε να ακούσουμε και περισσότερα σχετικά με τις τελευταίες νομοθετικές προτάσεις ε, για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων και για το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας γιατί και αυτό είναι στο πεδίο αρμοδιοτήτων του κυρίου Μοέντας. Τρία ζητήματα λοιπόν. Η σύγκριση του πρόγραμματος Πλησίου 9 με τον ορίζοντα 2020, η σημερινή κατάσταση στο ορίζοντα 2020, τα προγράμματα εργασίας 2018 ως 2020 και το πρόγραμμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε και κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, όπως πάντα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή στιγμή για ανταλλαγή απόψεων και θα με βοηθήσει στην καθημερινή μου εργασία. Να πω δύο λόγια για τα τελευταία τρία χρόνια, για το παρόν και το μέλλον. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρία χρόνια που πέρασαν. Νομίζω ότι περισσότεροι έχετε λάβει μέσω email ε, το φυλάδιο για τα τρία χρόνια του ορίζοντα 2020. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιους αριθμούς ε, που είδατε εκεί μέσα για το τι έχει γίνει. Έχουμε λάβει πάνω από 150.000 επιλέξιμες προτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν δείτε τις προτάσεις ε, υψηλής ποιότητας δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε ε, πολύ καλά επιστημονικά προγράμματα. Νομίζω ότι οι υπολογισμοί είναι απλοί. Με τον τωρινό προπολογισμό μπορούμε να στηρίξουμε μόνο μία στις τέσσερις προτάσεις. Οπότε παραμένουμε ελκυστικοί, αλλά είμαστε θύμα της επιτυχίας μας, θα έλεγα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, είναι να πείσουμε τις ε, χώρες Και βεβαίως ε, χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά για το μέλλον. Αν δείτε λοιπόν ε, το ποσοστό επιτυχίας σε σύγκριση με το πρόγραμμα 7 που ήταν πάνω από 12% τώρα έχει πέσει στο το 18% έχει πέσει στο 12,6%. Τα βλέπει ο κόσμος και λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και ε, ναι, πράγματι υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έχουμε αρκετά λεφτά να χρηματοδοτήσουμε τα επιτυχή προγράμματα. Ο μέσος χρόνος επιχορήγησης έχει βελτιωθεί πολύ και αυτό νομίζω οφείλεται στην δουλειά των υπηρεσιών. Μιλάμε για 111 ημέρες πιο γρήγορα από ότι στο πρόγραμμα πλαίσιο 7. 90% δηλαδή των ε, συμφωνιών έχουν υπογραφεί μέσα σε 8 μήνες, αλλά η πιο θετική είδηση, θα έλεγα, των τριών ετών είναι ότι όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα με ρωτήσατε για το πώς ε, θα είναι ανοιχτό αυτό το πρόγραμμα σε νέους ανθρώπους ε, και σε νέους συμμετέχοντες και χαιρόμαστε πολύ για το ότι στα τρία αυτά χρόνια πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες είναι νέοι συμμετέχοντες, δεν είχαν έρθει στο πρόγραμμα πριν και είχαν τώρα την δυνατότητα να ενταχθούν. Αν δείτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, βλέπετε τα ίδια θετικά αποτελέσματα. 25,4% της χρηματοδότησής μας ε, που αφορά κυρίως ε, τα θέματα τεχνολογικής ηγεσία και κοινωνικών προκλήσεων είναι πάνω από το 23% που είχαμε ξεκινήσει. Αν δούμε όμως την κατανομή, γιατί τα τρία αυτά χρόνια μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια ευρώ, Βλέπουμε ότι 20% αυτών, το 1 πέμπτο, είχε πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Αλλά για να έχετε μια ιδέα, 20% του προϋπολογισμού πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. 40% του προϋπολογισμού πήγαινε για κοινωνικές προκλήσεις βασικά δηλαδή στέγαση, ενέργεια, μεταφορές, ε, διατροφή, περιβαλλοντικά. Και ο στόχος που είχαμε 60% δηλαδή ε, της χρηματοδότησης να αφορά βιωσιμότητα κτλ. επετεύχθη. Οπότε υποστηρίζουμε ολόκληρη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας από την βασική έρευνα μέχρι την καινοτομία. Μετά ενδιαφέρον να δούμε τις χώρες και το ποιες ε, είναι αυτές που ανταγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο. Βλέπετε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Γερμανία είναι στις πρώτες θέσεις, αλλά αυξάνεται κάθε χρόνο η συμμετοχή και είναι καλύτερη κατάσταση από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αυτός είναι και βασικός μας στόχος. Ποιοι είναι λοιπόν οι δικαιούχοι. 40% είναι πανεπιστήμια, κατά το οποίο δείχνει ότι είμαστε δυνατοί στα πανεπιστήμια, βιομηχανία 30% και ερευνητικά κέντρα ε, γύρω στο 8%. Επίσης να τονίσω το θέμα της ισορροπίας των φύλων. Το παλεύουμε και έχουμε πετύχει 55% των, της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής να είναι γυναίκες και 40% των ειδικών στα πάνελ αξιολόγηση να είναι γυναίκες. Αν αρκεί αυτό, όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ειδικά στα πάνελ νομίζω ότι εκεί είμαστε στο 40% πρέπει να ανέβει το ποσοστό αυτό και θα συνεχίσουμε βεβαίως σε αυτό το μέτωπο. Δεύτερον, το παρόν. Τι κάνουμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε μια ανακοίνωση για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν δύο βασικά σημεία εκεί. Το ένα ήταν η έκθεση την οποία όλοι γνωρίζουμε και το άλλο ήταν η πολύ σημαντική συνεισφορά της έκθεσης ε, Σαν Λουίς ε, Αυτά νομίζω ήταν τα βασικά σημεία αυτής της αξιολόγησης και σας ευχαριστώ. Και εάν δούμε τα διδάγματα που αντλήσαμε από αυτά, εγώ θα έβλεπα τρία σημαντικά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα η υψηλή προσθέμενη αξία. Ε, και σήμερα ακόμα βλέπω συζητήσεις ε, σε κάποιες χώρες για την προσθέμενη αξία του ορίζοντα 2020. Η προσθέμενη αξία είναι ξεκάθαρη. Στο 83% των έργων ε, το ποσοστό αυτό δεν θα είχε γίνει χωρίς ε, τον ορίζοντα 2020. Το 80% των έργων δεν θα είχε γίνει. Ε, και πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Δεύτερον, η χρηματοδότηση. Και εδώ πέρα η έκθεση, η Λανή και η Κάμπος Ανρίς οι εκθέσεις αυτές είναι ξεκάθαρες και στις είπα ότι και αν μας αρέσει, αν μας αρέσει η τωρινή ηγεσία στις είπα εξακολουθούν να επενδύουν 150 δισεκατομμύρια περισσότερα από εμάς. Αυτό είναι το γεγονός. Τρίτον, θεωρώ ότι και οι δύο εκθέσεις και η ενδιάμεση έκθεση νομίζω αντλεί το δίδαγμα ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινή προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω και το από πάνω προς τα κάτω είναι να έχουμε αυτές τις ε, ιδέες και να έχουμε ε, επιστημονική έρευνα που θα πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη αποστολή και η σκοπιά από κάτω προς τα πάνω είναι το θέμα της καινοτομίας. Αν δείτε λοιπόν αυτά τα διδάγματα και το έχουμε δει νομίζω στο πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 ξεκινήσαμε το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα με το μέσο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα κάναμε την πρώτη δημοσκόπηση όπου δεν υπάρχει θέμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 10 Ιανουαρίου. Λάβαμε πάνω από χίλιες προτάσεις για, το, για την πιλωτική διάσταση, οπότε έχουμε την πλευρά της ζήτησης του πιλωτικού σκέλους ε, και έτσι ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και το μέλλον είναι το προγραμμα εργασια εργασίας 2018-2020. Το παρελθόν, στο παρελθόν ήταν γύρω στα 25 δισεκατομμύρια και για τρία χρόνια και τώρα έχουμε γύρω στα 30 δισεκατομμύρια το 2018 μέχρι το 2020. Ποια είναι τα διδάγματα που προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα, να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και να απλοποιηθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα. Αυτά είναι πρώτα-πρώτα αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω για το πρόγραμμα 2018-2020. Η έκθεση να ρωτήσει, είναι ξεκάθαρη στο εξή. Έχουμε το θέμα της υπερεγγραφής με το να περνάμε σε μια διαδικασία δύο φάσεων και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πολλοί περνάνε στην πρώτη φάση, μετά περνάνε στη δεύτερη φάση, εξόδουν πολύ χρόνο και χρήμα και δεν φτάνουν στον τελικό. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον αριθμό ατόμων που περνάνε από την πρώτη στη δεύτερη φάση και να έχουμε μία λύση για ένα πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο δικαίω. Επίσης ε, τώρα περάσαμε και στις προκηρύξεις ε, του ποσού κατά Έχουμε δύο είδη προκηρύξεων και πολλοί μου είχατε πει σε διμερείς επαφές γιατί να μην έχουμε μία χρηματοδότηση κατά αποκοπήν. Να έχει ο κόσμος ε, ένα στόχο, τον πετυχαίνει και του δίνουμε τα λεφτά. Μετά έχουμε τα βήματα για να χρηματοδοτηθεί η πιλωτική φάση και μετά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, για την στήριξή σας και μετά πρέπει να γίνουν κάπως πιο λογικές οι προτεραιότητες. Έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες. Το κλίμα και ο άνθρακας 3,3 δις, κυκλική οικονομία 1 δισεκατομμύριο, ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 1,6 δισεκατομμύρια, η Ένωση Ασφαλείας με 1 δισεκατομμύριο και ακόμα και αυτά τα οποία δεν είναι ε, σε αυτές τις τέσσερις ε, προτεραιότητες ε, Έχουμε τα θέματα που μας απασχολούν, όπως η μετανάστευση που θα απασχολήσει πολλούς τομείς ε, και είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και έτσι έρχομαι στα τελευταία δύο σημεία. Το πρόγραμμα πλαίσιο 9 και όσα έχω πει τα τρία χρόνια αυτά για το πώς ενσωματώνουμε το πρόγραμμα εργασίας για το 18-20 και ποιοι είναι οι στόχοι μας. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι μελλοντικές ιδέες και στρατηγικές και πραγματικά μου αρέσει το όνομα αυτό, ορίζοντας κτλ. Και ήρθα για την συζήτηση σήμερα, αλλά και για να κάνουμε για μια και μια συζήτηση περισσότερο για το μέλλον. Πρέπει και αυτό να το δούμε. Κοιτώντας λοιπόν το πρόγραμμα πλαίσιο 9, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα. Πρώτον, κάτι το οποίο συζήτησα με τον πρόεδρο, τον Γκέρζι Μπούζεκ, για το χρονοδιάγραμμα. Και με ρώτησε μόλις ο πρόεδρος, είστε έτοιμοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Οι υπηρεσίες μας είναι έτοιμες. Βεβαίως, εξαρτάται από μας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Η έγκριση του ΠΔΠ και αυτό βεβαίω εξαρτάται από ολόκληρη την Κομισιόν και ειδικά τον κύριο Έτιγκερ. Αλλά μόλις εγκριθεί, εμείς είμαστε έτοιμοι. Μόλις εγκριθεί το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντα βεβαίως στα πλαίσια των κανόνων αλλά νομίζω μιλάμε για τον Μάιο περίπου, τα έχει πει ο συνάδελφος. Ε, είχαν καθυστερήσει οι συζητήσει και βεβαίω εδώ πέρα θα ακολουθήσω αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρο. Το πρόγραμμα πλαίσιο 9 θα είναι νομοθετικό πακέτο με πέντε τμήματα όπω το, το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν μία ανακοίνωση γενική, το πρόγραμμα πλαίσιο το ίδιο, το συγκεκριμένα πρόγραμματα και του κανόνε συμμετοχή θα υπάρχει μια ξεχωριστή πρόταση για την ευρατόμο συνήθως, και νομίζω ότι εάν δείτε τώρα το περιεχόμενο, το είχα περιγράψει στο παρελθόν ως αριστεία, αντίκτυπος ε, και ε, ένα πρόγραμμα ανοιχτό προς τα έξω και ακριβώς ε, το θέμα είναι πώς θα πάμε σε κάτι το συγκεκριμένο. Και μπορώ να σας πω το εξή. Ε, βεβαίως ίσως κάποιοι το έχετε ξανακούσει. Το πρόγραμμα αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη, όχι μια επανάσταση. Υπάρχει συνέχεια, συνέχεια στα πράγματα τα οποία κάνουμε καλά. θεμελιώδη, βασική επιστήμη. Δεν βλέπω κάποιε ιδιαίτερε αλλαγέ εδώ. Πρωτογενής έρευνα δηλαδή, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, ε, με τις δράσεις ε, Marie Curie και μετά έχουμε νέο τρόπο σκέψης, πώ θα σκεφτούμε διαφορετικά για το μέλλον και το πώς θα περάσουμε από τι κοινωνικές προκλήσεις, τι παγκόσμιες προκλήσεις, οι οποίες για εμένα είναι αυτές, αυτή η προσέγγιση η οποία είναι από πάνω προς τα κάτω και μετά υπάρχει ο τρίτος πυλώνας που αφορά την ανοιχτή καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Έχουμε λοιπόν θεμελιώδη έρευνα από πάνω προς τα κάτω, το Συμβούλιο καινοτομία και μετά έχουμε μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που δίνουμε κατευθύνσεις. Έχουμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι καινούργια, αλλά δεν είναι κάτι το επαναστατικό, είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή η ιδέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομία που έχουμε συζητήσει εδώ τόσο πολύ και κοιτάμε τώρα το, την πιλωτική φάση, να έχουμε συνεντεύξεις με τους επενδυτές, να έχουν περισσότερες δυνατότητες να προτείνουν ιδέες, να μην υπάρχουν θεματικοί περιορισμοί, να δημιουργήσουμε ακριβώς ε, τους καταλόγους αυτούς ε, των ε, ειδικών, των αξιολογητών. Δηλαδή τον έχουμε πάνω από 100 άτομα τα οποία θα είναι και επιχειρηματίε και μπορούν να δουν τα πράγματα με μία άλλη σκοπιά και να τα αξιολογήσουν. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό και τους ο κόσμο. και δεν επειδή ακούτε για πρώτη φορά αρχηγού κρατών όπω τον πρόεδρο Μακρόν να μιλάνε για καινοτομία ε, ή επειδή είναι τη ε, μοδός ε, επειδή σε τελική ανάλυση κοιτάω το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ποιο είναι το θετικό μήνυμα. Το θετικό μήνυμα είστε ε, εσείς η, η καινοτομία, η επιστήμη. Οτιδήποτε, για οτιδήποτε μιλάμε, από τρομοκρατία μέχρι πρόσφυγες, δεν είναι το θετικό μήνυμα. Είναι προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά το θετικό μήνυμα είναι, νομίζω, η δουλειά που κάνετε εσείς εδώ. Γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινοτομίας. Αλλά δεν αρκεί, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ακριβώς αυτές τις αποστολές για να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος το τι θέλουμε. Νομίζω ότι σήμερα εμείς ξέρουμε τι θέλει ο κόσμος, οι επιστήμονες μας καταλαβαίνουν, αλλά ο κόσμος απλώς δεν μας καταλαβαίνει. Γι' αυτό οι αποστολές ε, έχουν σημασία να έχουμε κάποιες ιδέες που ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, ο χρόνος πιέζει. Ε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλοι γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα που θα είναι πολύ δύσκολο και γνωρίζουμε επίσης ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά για να προετοιμάσουμε το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Λοιπόν, είναι προετοιμασμένες οι υπηρεσίες μου και εγώ θα σας βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Για εμένα λοιπόν το θέμα είναι αυτό ότι εμεί θέλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σε αυτή την θητεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, στην ε, δική σας θητεία. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Σας ευχαριστούμε για όλες τις ε, πληροφορίες για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Αναφερθήκατε σε δύο χαρακτηριστικά που δεν είναι επαναστατικά κτλ. Θα ήθελα να προτείνω η συζήτηση μαζί σας, αγαπητά μέλη, να γίνει ως εξή. Καταρχήν, να πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, οι επίσημοι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, για τρία λεπτά το πολύ. Σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεύτερον, για δύο λεπτά οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές ε, για την εφαρμογή την έκθεση εφαρμογή του προγράμματο Οριζόντα 2020 και κατά τα άλλα οι λοιποί ομιλητέ για ένα λεπτό. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε αρκετό χρόνο για μακροσκελή συζήτηση. Να περάσουμε λοιπόν στου προσώπου των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Έλερ, εκ μέρου του ΕΛΚ. Τρία λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους. Ε, όταν ε, έχει κάποιο στη θέση τρία λεπτά, φυσικά δεν μπορεί να καλύψει πλήρως το πρόγραμμα. Αλλά θέλω να πω ότι σε 19 ομάδε εργασία, όπου συζητούσαμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη το θέμα τη ενδιάμεση αξιολόγηση, μπορώ να πω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά από αρκετού συναδέλφου. Θέλω να αναφερθώ στο ποιε ήταν οι φιλοδοξίε και τα ενδιαφέροντα του Κοινοβουλίου στο παρελθόν. Νομίζω ότι η ιδέα του fast track και το από κάτω προς τα πάνω ακολουθεί σε δύο κατευθύνσεις. Καταρχήν ότι θα πρέπει να είναι πιο ταχύ το πρόγραμμα, ακριβώς επειδή αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της παγκοσμίας οικονομίας, ε, αλλά και του ερευνητικού κόσμου. Μέχρι τώρα είχαμε πιλωτικό στάδιο, ε, τώρα έχει κατανεμηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνάς. Ε, όμως ε, πρέπει να δούμε και ποια είναι η εντύπωση από το πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο. Τώρα για την απλούστευση υπάρχει μεγάλη αναφορά στους ελέγχους δυνάμει επιδόσεων κτλ όντω ε, να πάμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ποιε είναι οι ικανότητέ μα. Ε, έχουμε μέχρι τώρα 50 ελέγχου ε, και κανένας δεν έχει βασιστεί σε δείκτες επιδόσεων. Το μόνο που έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο είναι για το γιατί. Έτσι λοιπόν, πώς, πόσο ρεαλιστικό είναι να αλλάξει το σύστημα. Τρίτον, για την αποστολή. Συμφωνώ με την ιδέα και τη χαιρετίζω, αλλά θέλω να αναφερθώ στο σκέλος του προγράμματος Επιστήμη και Κοινωνία. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος ε, για να υπάρχει αποδοχή του προγράμματος και τι θα γίνει με αυτό. Θέλω να αναφερθώ και στο ΕΡΑ, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Έχουμε ε, ουσιαστικά κάποια τμήματα του προγράμματος που είναι πιο απομονωμένες ε, και τι θα γίνει, θα ενταχθεί ή εξακολουθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας να αποτελεί ένα όνειρο και υπάρχει και το θέμα τη ανοιχτή πρόσβαση. Βλέπουμε τη φιλοδοξία, μιλάμε συνέχεια για ανοιχτό χαρακτήρα, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε σύστημα δημοσίευση και αν θέλουμε να δημοσιεύουμε τα πάντα, ρεαλιστικά δεν υπάρχει ε, ουσιαστικά κανένα σύστημα διορισμού για ένα καθηγητή που να βασίζεται σε μια ανοιχτή διαδικασία. Αν θες να γίνεις καθηγητής ε, πρέπει να δημοσιεύεις και ο ρυθμός των δημοσιεύσεων κρίνει αν θα διοριστείς. Έτσι λοιπόν μιλάμε για γενικό χαρακτήρα, είναι πραγματικότητα για ένα καθηγητή είναι ότι δεν έχει νόημα για ανοιχτή πρόσβαση γιατί ακριβώς διορίζεται επειδή δημοσιεύει, κάνει δημοσιεύσεις. Σε σχέση λοιπόν με το ΕΡΑ, μήπως ε, αυτό το ανοιχτό ε, θα αποτύχει αν δεν το μεταφράσουμε σε εθνικά προγράμματα και για τις συνέργειες ε, κάτι τελευταίο. Θέλουμε να έχουμε τη γέφυρα με το διαφορετικό τομείο, αλλά έχουμε αυτό το λευκό ελέφαντα στο δωμάτιο. Και ουσιαστικά, τι λέμε, είναι ουσιαστικά πρακτικό λόγο της κρατικής ενίσχυσης δεν ε, θα πρέπει ίσως ε, στο μέλλον ε, να μιλάμε για συνέργειες, αλλά πρέπει να βρούμε ακριβώς απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Η κυρία Καμπεσον από τους Σοσιαλιστές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πίτροπε. Καταρχήν, να σας πω ότι χαίρομαι που τελικά δημοσιεύτηκε αυτή η ανακοίνωση και μπορούμε να συντονιστούμε. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν να συντονιστούμε για το έργο που απαιτεί το επόμενο πρόγραμμα. Έχουμε σημειώσει σημαντική δουλειά και θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε. Και από ό,τι φαίνεται τελικά μπορεί να ελοπιθεί αυτό. Εσείς ε, μιλήσατε για την συνέχεια, όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για προβλεψιμότητα ε, σε σχέση με το πέρασμα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το πρόγραμμα παρά τα καλά αποτελέσματά του. Και το τελευταίο γενικό σχόλιο είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνένεση που υπήρχε εντός της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για να συνεχίσει να έχει την εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας ε, το πρόγραμμα. Εμείς πρέπει να εργαστούμε για να το πετύχουμε εκ νέου στο πρόγραμμα αυτό. Και πιο συγκεκριμένα να πω ότι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία μετράται ε, ως προς ε, το μέγεθος της συμμετοχής, αλλά πρέπει να δούμε και πώ μετράμε το πραγματικό, τον κοινωνικό αντίκτυπο, πώς τα αποτελέσματα φτάνουν στην κοινωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να εργαστούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι πρόκληση να ξέρουμε ήδη πώ να το μετράμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από συγκεκριμένους ή πιο ευέστερο τομέα, όπω η πιο ευαισθητου τομει οπω η υγεια Ω προ την ε, δομή. Εγώ νομίζω ότι λειτουργεί η δομή, λειτουργεί καλά. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη συμμετοχή των κρατών μελών ε, και της βιομηχανίας. Είναι σημαντικός ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τον αυξήσουμε, αλλά δεν αρκεί για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε παγκοσμίω ε, σε θέματα έρευνας και κοινοτομίας. Θα πρέπει να δούμε πώς δεσμεύονται τα κράτη-μέλη και να κάνει και μια προσθέμενη προσπάθεια η βιομηχανία. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση αλλά και για την πρόταση του επόμενου προγράμματο ε, θα ήθελα να μιλήσουμε για τον κοινωνικό αντίκτυπο, όχι μόνο να μιλάμε με όρου ανταγωνιστικότητα αλλά και για το πώς τα δημόσια κονδύλια θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης, να βρούμε στρατηγικές ε, για να καλύψουμε το χάσμα των φύλων. Επίσης, νομίζω πρέπει να εργαστούμε για το θέμα της κοινωνικής επιστήμης και δεν έχω δει και καμία πρόταση ε, για το πώς ε, θα εναρμονίσουμε τις κρατικές ενισχύσεις που αποτελούν εμπόδιο για τις συνέργειες. Θα πρέπει να ε, βρούμε πώς ε, τα δεδομένα θα πολλαπλασιάσουν την επιστήμη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε το χάσμα που υπάρχει ως προς τη συμμετοχή ε, μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Θα πρέπει να δούμε πώς όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάσουν αυτή την αριστεία και χρειαζόμαστε περισσότερα κέντρα αριστεία. Για το GTI υπάρχει μια πρόταση για το νέο GTI, για την ε, κοινοπραξία. Μιλούσαμε για την ανάγκη συνοχής. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να αναλύσουμε πώς λειτουργεί το GTI και για ε, το GTI λέγεται ότι έχει πολύ υψηλή αξία η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία. Όμως θα πρέπει να βελτιώσουμε την διαφάνεια στην κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία στο GTI. Τέλος, να σας ε, πω ότι ε, καλό είναι να βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, όμως ε, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Χρειαζόμαστε να εμπλέξουμε και την εκπαίδευση. Και αυτό από τα πρώτα βήματα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία στους νέους και πρέπει να δώσουμε μία όθηση στην καινοτομία και χρειαζόμαστε καλύτερη σύνδεση όχι μόνο με τα πανεπιστήμια αλλά και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικότερα. Και κάτι τελευταίο. Συγγνώμη, απλώς να σας πω για το πρόγραμμα 18-2020. Έχουμε την πρόκληση της ε, αντίστασης της ανθεκτικότητας στα μικρόβια. Χιλιάδες άνθρωποι ε, θα πεθάνουν λόγω αυτής ε, αυτή τη πρόκληση. Επομένω, πρέπει να κάνουμε κάτι. Εκ μέρου του ECR, ο κ. Χέλτερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν αναφέρατε το επόμενο βήμα. Ε, γιατί όχι ορίζοντας 2030. Αλλά θα ήθελα να κάνω, νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα που έχει η οικονομία που καθοδηγείται από την αγορά είναι ότι τα στελέχη ορίζεται όπως και όλοι μας ότι ο προϋπολογισμός για τον οποίο είστε εσείς αρμόδιος είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού Και εδώ έχω κάποια σχόλια και τρεις ερωτήσεις. Είναι προφανές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο... ε, και τώρα για το μέλλον όσον αφορά είτε ε, και τώρα για το μέλλον όσον αφορά αυτή τη συνάντηση κορυφής για την καινοτομία για την έρευνα την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια ψηφοφορία ιστορική σημασία για πρώτη φορά έχουμε αυτό το μηδενικό στόχο για το 2050 στην Ευρώπη για ε, να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια ε, και για αεροπορικές μεταφορές και για θαλάσσιες και για τη χημεία για την ε, βιομηχανία γενικότερα αλλά για τις πόλεις τη σχέση και οικονομίας να εργαστούμε με τα κινήματα των πολιτών για να φτάσουμε σε αυτές τις μηδενικές ε, στο μηδενικό άνθρακα τέλο πάντων. Και εδώ θα πετύχουμε τη συνένεση εάν ασχοληθούμε πρέπει εκεί να δουλέψουμε σκληρά γιατί εκεί η επιστήμη δεν έχει προχωρήσει αρκετά πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόοδος εκεί ακόμα και με τις δεδομένες μεθόδους παραγωγής της βιομηχανίας. Άρα είναι θέμα τεχνολογίας, αλλά είναι και κοινωνικό. Άρα αυτό θα είναι πυρήνες σημαντικός ε, για την έρευνα. Τώρα κάτι άλλο. Πώς Μα τι θα, θα, θα, κάνουν, θα δώσουν τίποτα αυτοί οι ποινικοί δραστήρε σε 100 χρόνια. Θα είναι τελείω αποκεντρωμένο το σύστημα για αυτή την ε, σύνδεξη. Ε, θα είναι όλο ένα και... Χρησιμοποιήσουμε ε, ουσιαστικά τα κονδύλια για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Μπορέιλα, μου δώστε έξι λεπτά. Θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. δούμε την ενδιάμεση αξιολόγηση, κυρίως όταν βλέπουμε πόση επιτυχία έχει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε την ενδιάμεση αξιολόγηση και τα διδάγματα την προστιθέμενη αξία που προέκυψε από τον ορίζοντα 2020, τον αριθμό των ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου, προκειμένου να προσπαθήσετε να διασφαλίσετε ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 από την πλευρά τρίτων χωρών ε, είναι κάτι που έχει μία ακρόαση μαζί με τη ΣΤΟΑ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μείνει στις προτεραιότητές μας. Ναι, στην κυρία Κούτριτσκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε τον λόγο. Έχουν δύο άλλοι ομιλητές. Τώρα Εάν μου επιτρέπετε αγαπητοί συνάδελφοι, μην μιλήσετε περισσότερο από ένα λεπτό. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλουμε να μιλήσει και ο κύριος Επίτροπος. Και για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας θα είναι δύσκολο. Και πρέπει να τοποθετηθεί και ο ίδιος ίδιος. Κύριε Ζουρίνιο. Ευχαριστώ. Σα μία έντονη επιτάχυνση στην αναγκαιότητα έρευνα και κοινοτομία. Ε, είχα πάρα πολλέ ερωτήσει να θέσω, αλλά έχω μόνο ένα λεπτό. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας και να ρωτήσω ποιο είναι το όραμά σας για το πώς θα συνδυάσουμε τη σύγκληση με την του νέου προγράμματος εργασίας Δηλαδή, ε, όχι μόνο να λάβετε υπόψη αυτές ε, τις τρεις αρχές, την αριστεία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Η κυρία Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σε συγκεκριμένο πλαίσιο θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρόκειται για μια νέα έννοια, όλοι το γνωρίζουμε, όμως ε, λόγω ε, των ε, μαζικών σετ δεδομένων τίθενται πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει μια τεχνική συνιστόσα στον τομέα αυτό. Ε, τίθενται πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει μια τεχνική συνιστόσα στον τομέα αυτό. Όμως υπό την έννοια αυτή η καινοτομία είναι και οντολογίας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, βλέπει, σε ποιους τομείς ε, σχετικούς με την έρευνα βλέπει η Κομισιόν να αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και ποιος θα ήταν ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει στο μέλλον ο τομέας αυτός. Ευχαριστώ, κυρία Μάισνερ. η ωκεανή είναι πάρα πολύ σημαντική για το κλίμα, για την παραγωγή και τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα και ήδη έχουμε κάνει κάποια έρευνα στη θάλασσα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό για την εικόνα μας, αλλά και για την επιβολή μιας παγκοσμίας λύσης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπίρκουνεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας και για το υλικό που λάβαμε. Μας βοηθούν πάρα πολύ όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίαση του νέου προγράμματος πλαισίου 9. Νομίζω ότι η πυλώνηση είναι πολύ καλή, ε, χαρακτήρα χαρακτήρας ε, στην καινοτομία και στην ε, έρευνα, κλιματική αλλαγή κτλ. Και είναι πολύ σημαντικό και που επικεντρωνόμαστε και στην αριστεία ως προς τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Όμως, μια μεγάλη πρόκληση ήταν το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας ε, στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Τι μπορεί να κάνουμε τα επόμενα τρία χρόνια αν δεν πάρουμε τα πρόσθετα 70 δισεκατομμύρια για το πρόγραμμα. Τι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητέ μας γιατί κάνουν ε, πολλή δουλειά με τις προτάσεις τους. Και φυσικά δεν είναι πολύ ενθερητικό αν είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό επιτυχίας. Και θα ήθελα να μου πείτε και ποια είναι η άποψή σας για το Brexit, γιατί γνωρίζουμε ε, πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος του ΕΒ στον τομέα της έρευνας ε, και της κοινοτομία. Και ε, τώρα φαίνεται να σκοπεύει να σχεδιάσει ένα νέο να σχεδιάσετε ένα νέο πρόγραμμα και δεν ξέρουμε τι ποσοστό συμμετοχή να περιμένουμε στο μέλλον από το Ηνωμένο Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σμαρτέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, Επίτροπε εξαρτάται από το ΣΕΦΠ αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Γιατί αυτή η πρόταση κινδυνεύει να έρθει πάρα πολύ αργά. Και ε, τότε να περιμένετε την επόμενη θητεία. Επομένως ε, το μήνυμα παίρνουμε είναι κινδυνεύει να έρθει πάρα πολύ αργά. Και ε, τότε να περιμένετε την επόμενη θητεία. Επομένως το μήνυμα παίρνουμε είναι ευχαριστούμε πολύ κύριος Ρομπίχινο επόμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το φυλάδιο. Παρακαλούσα στο μέλλον να υπάρχει και ένας κωδικός QR, να το βλέπουμε σε ηλεκτρονική μορφή. Θεωρώ ο κόσμος ότι αυτό είναι το σημαντικότερο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία διαφορετικών ε, θεσμικών οργάνων και θα πρέπει ακριβώς να την μετράμε, να δούμε πώς αναπτύσσεται. Οπότε νομίζω να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός και το θέμα είναι τι θα γίνει με την έρευνα των υδάτων. Που μίλησα για το Brexit σχέση με το Horizon 2020 ε, είναι σκληρό το Brexit. Λέγεται ότι θα ωφεληθούμε από το Horizon 2020, αλλά επίσης είπατε ότι και η Ευρώπη ωφελείται από τη συμμετοχή της χρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Ε, φτιάξαμε ένα υλικό που παντού και σε υγεία, ε, χαμηλές εκπομπές διοξιδίου, σε ψηφιακά έχουμε ε, προχωρήσει εγώ συνεχίζω και ρωτάω τι αμοιβία σχέση μεταξύ έρευνας ε, καινοτομία στην ε, Βρετανία και τις αντίστοιχες προσπάθειες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ τα για αυτά. Το οποίο είπες, λέει πρώτος, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπες. Ο κύριος Κοχλίτσεκ έχει τώρα το λόγο. Για εμπλέκεται τόσο πολύ όσο το Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε στο περιθώριο ο κύριος ε, Τούρμες είπε ότι είναι αποκριστικό το ότι ε, το ΙΤΕΡ μπορεί να δημιουργήσει μία ε, συγκεντρωμένη πηγή ενέργειας να θερμάνουν έναν φούρνο κεραμικών. Οπότε χρειάζονται οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε ενέργεια και τις πηγές της ενέργειας. Έχει σημασία για την ανθρωπότητα. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σημασία και το ανέφερε η κυρία Μάισνερ είναι η ωκεανή. του Ατλαντικού υπάρχει ένα νησί πλαστικού μεγαλύτερο από την Ουκρανία που εμποδίζει την φωτο Θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα απόβλητα, γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα απόβλητα, στα σκουπίδια, στους χιτά, πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Διασμό, την οποία συζητήσαμε χτες, πρέπει λοιπόν να συνδεθεί και το πρόγραμμα αυτό με την οδηγία. Ευχαριστώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για το φυλάδιο. Έχει πολλές πληροφορίες, ε, αλλά στην κατηγορία 4. Η τρομερά χαμηλή αριθμή επιτυχών αιτήσεων. Αυτό δείχνει ε, πόσο μεγάλη υποχρηματοδότηση έχει το πρόγραμμα έρευνας ε, και σας ευχαριστώ εγώ. Θα ήθελα να σας παρακινήσω λοιπόν να φέρετε το πλαίσιο. Γιατί Εάν ισχύει αυτό το οποίο είπαμε ότι η ευρωπαϊκή προστάμενη αξία του προγράμματος αυτού είναι τόσο μεγάλη, τότε βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση και πόσο χαμηλή είναι η χρηματοδότηση. Και ακούμε διάφορα επιχειρήματα πορτοφόλι, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε τις εισφορές των Ελπίζω, κύριε Επίτροπε, να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, γιατί συνολικά είχαμε περίπου 35 ερωτήσεις. Πολύ μεγάλος αριθμός. Τέλεια. Κανείς δεν θα λέγει ότι είναι λάθος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις ερωτήσεις αυτές. Ο Επίτροπος ε, και το γραφείο του ε, υποσχέθηκε να μας απαντήσει όλες τις ερωτήσεις γραπτός. Όμως τώρα, το πιο σημαντικό, τώρα δεν ξέρω, ίσως δεν είναι δυνατόν να επιλέξει κανείς, αλλά ας δώσουμε στον Επίτροπο το λόγο, ίσως ε, για 6-7 λεπτά και πάλι είναι αρκετός χρόνος, κύριε Επίτροπε, αλλά για 35 ερωτήσεις δεν είναι τίποτα, γιατί είναι 10 δευτερόλεπτα για μία ερώτηση. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Θυμηθείτε ότι θα απαντηθούν όλες ε, οι ερωτήσεις και οι αμφιβολίες σας γραπτός. Συμφωνήσαμε από αυτού. Και τώρα ας ακούσουμε τις τελικές σας παρατηρήσεις, παρακαλώ. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θα ξεκινήσω αμέσως. Ε. Κοιτάξτε, να αρχίσω και να απαντώ με τη σειρά. Καταρχήν για τον κύριο Έλερ σε σχέση με το ΕΣΥ έχουμε τώρα αυτά τα τρία δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο το χρόνο για την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αυτή την πρωτοβουλία. Για την ανοιχτή πρόσβαση πιστεύω ότι ε, ο τρόπος που κάθεσαν ε, οι Γερμανοί με 200 ε, πανεπιστήμια να συζητήσουν ε, για το θέμα των δημοσιεύσεων ε, και είπαν ότι πλέον δεν θα είμαστε πελάτες. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι και η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το συζήτησα με τους Γερμανούς Πριτάνης. Έτσι λοιπόν, για να απαντήσω τώρα στην κυρία Γκαμπέσον Ρουίς, πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας, συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να είμαστε καλύτεροι και όλα σχετίζονται με τον κοινωνικό αντίκτυπο, με την προβλεψιμότητα. Μιλήσατε και για τις κρατικές ενισχύσεις, τον ορίζοντα του 2020 και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και η κυρία Βίνκερ ε, με ρώτησε για την ε, ανθεκτικότητα στα μικρόβια, την μικροβιακή ανθεκτικότητα υπάρχει ένα άρθρο από τον καθηγητή Κούζενς στο Nature για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το θέμα της ανθεκτικότητας στα μικρόβια που θα πρέπει να το διαβάσετε. Γιατί όλα έχουν γίνει στην Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, για την αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα άλλαξε τα πάντα. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να το λύσει σε κρατικό επίπεδο και τα project που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πραγματικά μοναδικά. Τώρα, ο κύριο Σέγγελ ε, με ρώτησε, μου έθεσε μια πολιτική ερώτηση για το Brexit. Είναι μια κατάσταση την οποία χάνουν όλοι, ναι. Είναι απώλεια για όλους. Ε, νομίζω αυτό είναι το λυπηρό γεγονός. Ε, θα πρέπει να αγωνιστούμε όσο περισσότερο μπορούμε για μια μελλοντική σχέση με το Ερμένο Βασίλειο, με όρους έρευνα και καινοτομίας. Ναι, εγώ θα αγωνιστώ όσο μπορώ για να υπάρξει αυτή η σχέση, ακριβώς γιατί τους χρειαζόμαστε και μας χρειάζονται. Επίσης ρωτήσατε, είναι δυνατό να έχουμε μια σχέση όπως έχουμε την Ελβετία και το Ισραήλ. Δεν είναι συγκρίσιμο γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόνο μεγαλύτερο από αυτές τις χώρες και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, δεν εξαρτάται από μας ε, δυστυχώς ε, και απαντώ και την ε, άλλη ερώτηση που τέθηκε σχετικά. κυρία Βερίνκε έκανε ένα σχόλιο για την αριστεία. Ουσιαστικά αναφερθήκατε και στον θέμα των δύο σταδίων. Θα δούμε αυτά τα δύο στάδια στο επόμενο πρόγραμμα, πιο σωροποιημένα. Δεν θέλουμε να δαπανίσουμε χρήματα ή χρόνο. Αλλά υπήρχε και ερώτησή σας για τα διευθυντικά ταμεία. Νομίζω ότι άπαξα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα που κάναμε. Καλό, έχουμε ουσιαστικά κέντρα αριστείας και θα πρέπει ουσιαστικά να το επαναλάβουμε έτσι ώστε ε, να εργάζονται πάρα πολύ καλά παρόλα κάποια προβλήματα κρατικής ενίσχυσης που είχαμε. Αυτά τα κέντρα ε, αυτή η σφραγίδα αριστεία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι πήγαν στα διαφορετικά ταμεία και έλαβαν τα κονδύλια. Θα πρέπει να έχουμε μια αναλογία, αν δεν έχουμε τα χρήματα, να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν κονδύλια από τα διαφορετικά ταμεία. Και αυτή η συνέργεια είναι απαραίτητη. Ο κύριο Τουρμα δεν είναι εδώ. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε να συζητήσουμε διμερώς για αυτό το θέμα, γιατί ήταν μακρά η ερώτηση, μακροσκελής με όλα όσα είπατε ε, σε σχέση με το να έχουμε μεγαλύτερη κατανομή. Είναι πολύ μεγάλη πολιτική πρόκληση για τα επόμενα δέκα χρόνια για το πώς είναι αυτά ε, που ε, ουσιαστικά ε, συμμετέχουν. Εμείς δίνουμε κάποιες υποτροφές ε, τον αντίκτυπο με την αριστεία και με τον ενικό χαρακτήρα. Αυτοί οι όροι φυσικά συμπεριλαμβάνουν και το θέμα της σύγκλησης. Συγγνώμη, θα περάσω στα κυβερνήσεων. Αυτό είναι το κύριο θέμα μας εδώ. Θα πρέπει να βγούμε από αυτή την αίθουσα και να πάμε στους υπουργού Οικονομικών. Και ξέρω κάποιοι μερικές φορές απευθύνονται στους υπουργού Οικονομικών και είναι εξάρτητα από όλη την Ευρώπη θα υπάρξει ένα έγγραφο σε μία εβδομάδα όπου θα έχουμε μία ανεξαρτησία εδώ με την πρόταση για το πρόγραμμα πλαίσιο 9 και να σας πω ποιες είναι οι ακριβείς αποστολές. Όπως είπατε, πρέπει να έρθουμε με τα κριτήρια για αυτές τις αποστολές. Ε, Πιλέρ Δελκαστήγιο, σε σχέση με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό είναι το κύριο ζήτημα για το μέλλον πρέπει να λάβουμε καταρχήν μια πολιτική απόφαση. Έχει επίπτωση σε όλου του τομεί. Η κυρία Μέσνη ρώτησε για την ε, μπλε οικονομία, την γαλάζια οικονομία, του ωκεανού. Προκάτοχό μου την βιοοικονομία και δεν υπάρχουν στο φυλάδιο αυτά. Ζητώ συγγνώμη, θα επανέλθω και θα σας στείλω περισσότερες πληροφορίες. Ε, κυρία Βικόνεν, με ρώτησε για τον Brexit. Μαρτέν. Εγώ σκεφτόμαι ότι υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα, δηλαδή για το πολιτές δημοσίου. Χρειάζομαι τη δική σας βοήθεια, κύριε Ρούμπικ. για το θέμα της επικοινωνίας που νομίζω, το οποία οι άνθρωποι θα πούνε να καταλαβαίνουμε τι κάνουν αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες. Τερέσα, νομίζω ότι απάντησα κάπως στην ερώτησή σου. Είχε ε, βρει πως ένα βακτήριο ε, θα προστατεύσει από τη γρήπη και ουσιαστικά ήταν μία μυς. Και τέλος κύριε Γκάιερ, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και την υποστήριξή σας. Στο τι είπατε... Απίστευτο αγαπητοί φίλοι. 40 ερωτήσεις σε 10 λεπτά και ικανοποιηθήκατε οι περισσότεροι. Οι υπόλοιποι θα λάβετε απαντήσεις γραπτός, γιατί Κάποιες έμειναν απάντητες, τα πρόσεχα όλα. Τελευταία μου σύμβουλη, κύριε Επίτροπε, αν μου επιτρέπετε, τα τελευταία έργα του προγράμματος πλαισίου 9 θα τελειώσουν θα τελειώσουν ε, το 2030. Θα μπορούσε να δηλαδή ορίζοντας 2030. Με κάτι το επαναστατικό οπωσδήποτε. Το τελευταίο έργο θα τελειώσει αρχές του 30. 2030. Αν αποφασίσετε κάτι τέτοιο λοιπόν, να μην πάτε με την χρηματοδότηση, πηγαίνετε ένα έργο. Α, ε, θα δούμε βεβαίως, γιατί και το όνομα έχει σημασία. Ο ορίζοντας 2020 ήταν πολύ σημαντικό όνομα και από αυτήν την άποψη ε, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι προετοιμαζόμαστε για το 2020, όχι μόνο για την αυριανή ημέρα. Σας ευχαριστώ. Τώρα μια σύντομη ενημέρωση στο επόμενο σημείο, γιατί σε 2-3 λεπτάκια θα έρθει η κυρία Επίτροπος εδώ. Λοιπόν, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση. Ζητάμε συγγνώμη την κυρία Επίτροπο. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Συνάδελφοι, μια σύντομη πληροφορία. Κβαντική, ε, πρωτοβουλία κβαντικής τεχνολογίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Και παρουσίαση θα κάνει ο καθηγητής Μάζο Καλάρκο. Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, ε, γιατί δεν υπάρχει αρκετό χρόνος ε, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, γιατί είστε διευθυντής του Κέντρου Ολοκληρωμένης Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ούλμα. Και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε ε, και να ακούσουμε τα συμπεράσματά σας. Κύριε καθηγητά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτέ, κύριε και κύριοι, ε, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, αν και θα πρέπει να βιαστώ λίγο γιατί είχα προετοιμαστεί για περισσότερο χρόνο να πω ένα πράγμα για την κάθε διαφάνεια. Το σημαντικό θέμα λοιπόν εδώ πέρα είναι οι αποστολέ. Ε, όπως είπε και ο επίτροπο Μαμόδας, το θέμα είναι πώ θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με το κοινό. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι το εξή. Πλησιάζουμε ήδη στη μελλοντική εποχή κβαντιοτεχνολογία γιατί γνωρίζουμε ότι οι επεξεργαστές των πολιτών γίνονται όλο και μικρότεροι και πηγαίνουμε πλέον στο μέγεθος του ατόμου και ήδη βρισκόμαστε σε, στην φάση της πρώτης κβαντικής επανάστασης. Ναι, Έχουμε δηλαδή ε, συσκευές, ε, έχουμε πολλά δισεκατομμύρια ηλεκτρονίων, φωτονίων. Εδώ πέρα βλέπετε τον Δαλάη Λάμα όταν τον συνάντησα στο Ίνισμπρουκ όταν ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητή, είχε έρθει να δει κάτι το τελείως καινούριο. Η δυνατότητα, η καινούρια τότε, ε, να χειριστούμε, το οποίο ανοίγει βεβαίως τον δρόμο για νέες εφαρμογές. Να σου πω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ πέρα βλέπετε έναν δορυφόρο. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω ε, τις λεπτομέρειες ακριβώς ε, της ε, κβαντικής εμπλοκής η οποία απασχόλησε οι ασφαλείς επικοινωνίες. Αν στέλνουμε λοιπόν με μονομένες φωτογραφίες είναι αδύνατον κάποιος ε, να τις υποκλέψει χωρίς να το παρατηρήσουμε. Από τους νόμους της φυσικής λοιπόν καθίσταται αδύνατη η υποκλοπή. Από την άλλη, ένα από λίγες ε, ημέρες ε, στην έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών, ένα τσίπ, έναν μικροεπεξεργαστή κβαντομηχανικής, ο οποίος θα έχει εφαρμογή στην βελτιστοποίηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά θα υποστούν μια επανάσταση με μεμονωμένα Ο Κλασικός ε, υπερυπολογιστής, ο μεγαλύτερος τότε στην Ευρώπη και οι μπλε τελείες είναι αυτό το οποίο κάνει ένα κβαντικός υπολογιστής ο οποίος μετά δεν μπορεί να ακολουθήσει και περνάμε ένα κατόφλι πλέον ε, υπολογιστικής δύναμης για ε, παραδείγματος χάρη επηρεάζονται από το μαγνητικό πεδίο ενός νευρώνα στον εγκέφαλό σας. Θα το παρατηρήσει λοιπόν αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά πράγματα, για ιατρικέ διαγνώσεις, για την ε, ναυσιπλοεία, τα συστήματα, κατεύθυνση του αυτοκινήτου σα και τα λίστε Έχουμε πολύ ε, εξέχουσες ομάδες. Έχουμε πολλές εταιρείες που παρέχουν την σχετική τεχνολογία και πολλές νέες επιχειρήσεις στον τομέα αυτών. Κάθε φορά που πάω σε συνέδριο εμφανίζεται μια νέα εταιρεία, οπότε είναι δύσκολο να παρακολουθήσω τις μικρές αλλά και τις για να κάνει μια προσωμείωση της κίνησης των ταξί στο Πεκίνο, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και βλέπετε ακριβώς γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες εταιρείε που έχουν εμπλακεί στην διαδικασία την Bosch, Airbus, Atos, KPN, Ericsson κτλ. Εδώ πέρα στην Ευρώπη λοιπόν το θέμα αφορά με σημαντικά εθνικά προγράμματα με πάνω από 500-600 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων ήδη. Λοιπόν, ποια είναι η αποστολή μας. Κάτι το συμβολικό, όπως ο άνθρωπος που πήγε στο φεγγάρι, για να έχουμε του χάρη, περάσω τώρα τις τεχνικές λεπτομέρειες αν μου επιτρέπει ο πρόεδρος, και εδώ πέρα έχουμε τους τέσσερις τομείς που ανέφερα βασίζονται, όπως είπαμε, στην βασική έρευνα και χάρηκα για αυτά τα οποία άκουσα, γιατί έτσι ακριβώς μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία αύριο και μεθαύριο. Εδώ πέρα λοιπόν δεν υπάρχει χρόνος για Για το 2035 την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την ανάπτυξη μετά αυτών των τεχνολογιών. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ Ωραία, τι θα έλεγα, τεχνολογία και εδώ πέρα ο καθένας ε, μπορεί να... Εδώ πέρα έχουμε την έκθεση της Επιτροπής μας ε, που περιέχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες την οποία παραδώσαμε πριν από λίγους μήνες στον Αντιπρόεδρο σε Ελπίζω να ήμουν αρκετά γρήγορος. My goodness, professor, it is possible for... Μόνο αν κανείς τα καταλαβαίνει όλα και άλλα τόσα μπορεί να τα πει όλα σε έξι λεπτά. Γιατί αυτό αφορά τις εξελίξεις των επομένων δεκαετιών για το πώς θα χτίσουμε αυτά για το μέλλον και επίσης και βοσκοπεί και το ορίζον 2020. Οπότε αν εσείς συνάδελφοι και πολιτικές ομάδες αποφασίσετε ότι χρειάζεται να τα πούμε διαμακρών με τον καθηγητή και να τα συζητήσουμε ενδελεχέστερα. Όπως εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε εδώ τις ε, προτάσεις σας, τις διαφάνειές σας για να προετοιμαστούμε να τα συζητήσουμε και εμείς, να σας υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις γιατί σήμερα είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε να ξανασυναντηθούμε με τον καθηγητή, εάν συμφωνείτε εσείς βεβαίως. Ήταν τέλεια, ήταν πολύ σύντομο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. So, dear friends, ε, hot time. Αγαπητέ φίλοι, και τώρα ήρθε η ώρα. Ε, πολύ σημαντικό που για κάθε επιτροπή έχουμε εδώ την ε, κυρία Γκάμπριλ την Επίτροπο. Ελάτε. member of European Parliament. I understand very well. Um, well, uh, your batch will... Ξέρετε, ως πρώην Ευρωβουλευτής, θα είστε πρώην Ευρωβουλευτής και θα ισχύει η ταυτότητα ισχυρική που έχει πολύ περισσότερο από την ταυτότητα του Επιτρόπου. Οπότε μονάζει δικά σας και εγώ να σας πω ότι έχουμε αυτόν τον διαρθρωμένο διάλογο το δομημένο διάλογο που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε. Είναι το θέμα του νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλεια. Θεωρούμε ότι το θέμα μας αφορά 100% είναι δική μας αρμοδιότητα. Όπως έχει ε, κρυφθεί από το Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω ότι κάποια από τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας και Γκάμπριελ, τη τηλεπικοινωνία, η ασφάλεια, ε, είναι πολύ σημαντικά. Οπότε και αυτό και σας ε, παρακαλούμε να μας παρουσιάσετε αυτό το νομοθέτημα. Έχεις το λόγο, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, μέλη τη Ήτρα, πρώτα πρώτα σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα από τα θέματα προτεραιότητάς μου ως Επιτρόπη με το χαρτοφυλάκιο του ότι ήδη με έχουν εντυπωσιάσει οι γνώσεις σας επί του θέματος. Οπότε και σήμερα μπορούμε να επισέλθουμε κάπως στις λεπτομέρειες. είδαμε τη σχετική δέσμη μέτρων, ώστε να φτιάξουμε μια ανθεκτική ε, όσον αφορά τις απειλές ευρωπαϊκή. Και είπαμε για την Ίνσα ότι 80% των όσων ήταν στην διάσκεψη δεν ξέρανε για την Ενίσα. Τη δέσμη μέτρων κυβερνών ασφάλειας και πρώτα πρώτα θα ήθελα να σταθώ στην Ενίσα ότι από το 2005 η υπηρεσία αυτή έγινε προς ε, κρατημέλη και θεσμικά όργανα και ε, επομένως ε, αφετηρία την επιτυχία και έχουμε και κάποια διαρκή και ακριβέστερη εντολή για την υπηρεσία. Ε, καινοτομείο ήταν η θέση που δώσαμε έτσι. Θα μπορεί να παράσχει ε, την εμπειρογνωμοσύνη της όποτε χρειάζεται. Είναι αναγκαίο να έχετε αρμοδιότητες ε, στα πλαίσια της ε, διαδικασίας συνεργασίας για όλη την Ένωση, όποτε χρειάζεται, όποτε υπάρχουν κάποιες κρίσεις και διασυνοριακές τρόσων, οι πολίτες και οι τελικοί χρήστες να έχουν περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες και θα το κάνουν αυτό άπαξ και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αγορά και έτσι να υπάρχει εξοικονόμηση. στον τονίσω ότι το προτινόμενο πλαίσιο δεν οδηγεί σε κάποιο είδου άμεση υποχρέωση για τους πάροχους ή τους παρόχους υπηρεσιών με διάφορα συστήματα να προσαρμοστούν αυτά στις ανάγκες της αγοράς των μελών, διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας, ε, ούτως ώστε να μην έχουμε τάσεις για τα κυβερνώ. Οπότε αναβαθμίζω τώρα η Ένισα και με αυτή την πρόταση αλλά και στο Συμβούλιο γιατί θέλετε να προχωρήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος το συντομότερο των προτέρων Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε κυρία. Και τώρα, πρόσωπο των πολιτικών Αντίθεση της κυρίας Νίμπλερ, ο κύριος Πολορυμπήχη για το ΕΛΚ. Ναι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ την Επίτροπο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Η Ενίζα παίζει έναν ρόλο κλειδί μαζί με την Μπέρεκ γιατί χρειαζόμαστε την ενίσχυση και την και έτσι ώστε οι κρίσιμες υποδομές να παραμείνουν στο επίπεδο που χρειαζόμαστε σήμερα και στο μέλλον. Εξ ονόματος λοιπόν της Αγγέλικα Νίμπλερ να σας συγχαρώ για το σχετικό νομοθέτημα γιατί νομίζω ότι αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση συζήτηση Είναι η συγγήτρια της Επιτροπής μας και ζητά συγγνώμη σήμερα ε, γιατί όπως είπαμε κολλείται. Το βασικότερο θέμα λοιπόν είναι να το δούμε από την σκοπιά του καταναλωτή. Τι χρειάζεται ο καταναλωτής ε, και πώς μπορούμε να δώσουμε ακριβώς ε, την σωστή την εμπιστοσύνη που απαιτείται, ειδικά σε σχέση με το ίντερνετ των πραγμάτων. Εάν δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτό, βλέπουμε ότι η υποδομή, οι οπτικές ίνες ε, Ε, το γεγονός ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερα δεδομένα στο, περιβα... στο μέλλον σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και η ε, υποδομή αλλά και το απαραίτητο λογισμικό. Η Ευρώπη θέλει να παίξει ε, ηγετικό ρόλο στα συστήματα αυτά, στο μέλλον και στα συστήματα εμπιστοσύνης, στην κρίσιμη υποδομή. Όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία. Όσον αφορά το στο, πλαίσιο για την ενίσα, την υπηρεσία αυτή, υπάρχει ένα πλαίσιο πιστοποίησης ε, προϊόντων πληροφορικής, ε, το οποίο βεβαίω και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδιαμορφώσαμε. Και γεγονός είναι ότι έχουμε μια παγκόσμια ψηφιακή επανάσταση. Και γεγονός είναι ότι ε, τα δεδομένα μας είναι όλα ευάλωτα. Έχουμε την ε, κυβερνοκατασκοπία και το κυβερνοσομποτάζ που έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν ε, μια πιστοποίηση υψηλή ποιότητα, στο λεγόμενο σύστημα Trust και ακριβώς η εμπιστοσύνη είναι το βασικό ζήτημα στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε ως Ευρώπη κάποια αποτελέσματα και κάποια κράτη-μέλη ακόμα έχουν μείνει λίγο πίσω. Πρέπει να αναλύουμε προσεκτικά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την Ευρωπαϊκή Κυβερνοασφάλεια και τον ρόλο των κρατών μελών τον ρόλο που θα παίξουν τα καθοριστούν το πεδίο εφαρμογή ε, του σχεδίου που προτείνει η Κομισιόν εάν επαρκεί και αν είναι επαρκώς καθορισμένο. Για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ε, και το σχετικό κόστος ε, νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Τι γίνεται με καθαρίσουμε το εάν χρειαζόμαστε μία προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο ή αν θα έχουμε μια νέα προσέγγιση βιομηχανίας ε, το θέμα της πιστοποίησης, ε, τι μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα, πώς μπορούν να κλιμακωθούν σε μέγεθος αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μόνιμη έντολη, ο προϋπολογισμός, ε, το προσωπικό. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε την παγκοσμία Σενίζα είναι ακριβώς να δούμε το πώς θα υπάρξουν κάποιες όλα. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Αρκετά μεγάλη η ομιλία σας, ο κ. Κορουμπάτσεφ. Και τώρα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο και θα ήθελα να μιλήσω για τον τόπο της ΕΝΙΣΑ ως Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Χώρες όπως το Ισραήλ και η Σιγκαπούρη είναι μικρές σε μέγεθος, αλλά είναι πολύ προηγμένες σε αυτόν τον τομέα. Είστε και από τα 28 κράτη-μέλη. Είναι δυνατόν αυτό το πιστοποιητικό να συντονίζεται από την Κομισιόν ή από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά θα βοηθούσε αν αναγνωριζόταν και παγκοσμίω. Γιατί θα μπορούσε να προωθήσει Θα ήθελα να εκράσω τις ευχαρισίες μου για την προσέγγιση της Επιτρόπου, η οποία έχει προωθήσει ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Πριν 20 χρόνια δεν χρειαζόταν να προστατεύουμε τα τηλέφωνά μας και άλλες τέτοιες τεχνολογίες, ενώ είναι πολύ σημαντικός επαγγελματικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, ανησυχώ, μήπως η θα έπρεπε να είναι ε, η επαγγελματική οντότητα που θα συνεργάζεται με άλλους φορείς, όπως ο Μπέρ, κράτη μέλη. Βέβαια έχουμε την Europol ως έναν επιτυχή οργανισμό. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται με υπερβολικό άχθος για τη βιομηχανία. Αφενός θα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια ζωτική υποδομή και θα πρέπει να χαίρει πιστοποίηση, αλλά από την άλλη τα πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να γίνουν ένα είδος ε, αγαθού που θα είναι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και μεταξύ των ε, κρατών μελών να έχουμε ένα κεντρικό σημείο. Εγώ εκτιμώ αυτή τη δυναμική προσέγγιση που μας λέει ότι όλοι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ήδη πρέπει να τη χειριστούμε με ένα τρόπο ώστε να μην δημιουργηθούν μονοπόλια από κάποια κράτη-μέλη. Θέλω Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ράιμον για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο τις ερωτήσεις μας. Θεωρώ ότι οι τεχνικές εξελίξεις προχωράν πολύ πιο γρήγορα από τις πολιτικές εξελίξεις. Όταν ιδρύθηκε η ΕΝΙΖΑ δεν υπήρχε το Facebook. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι μιλάμε για πιστοποίηση σε ευρωπαϊκά κράτη και αμοιβαία αναγνώριση και βεβαίω καλό είναι να πατάμε ένα κουμπί και να φεύγουν τα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη σε πολλούς τεχνικούς χρήστες. Εν τω μεταξύ έχουμε την ελπίδα ότι θα μπλοκάρουν τα αμερικανικά κόμματα το ένα το άλλο και δεν θα υπάρξει ε, τελικά πρόοδο στη Βίζα, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Ο Τραμπ υπέγραψε μία παράταση κατά έξι έτη και όλα τα δεδομένα θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ για να τα παρακολουθούν οι εκεί μυστικές υπηρεσίες ε, και εντωμεταξύ τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια παρατηρήσαμε ότι και η Ρωσία κάνει hacking και το χρησιμοποιεί και πολιτικά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα κάνετε εσείς ως κομισιόν έτσι ώστε να δούμε το θέμα της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο πολιτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε για την παρουσίασή σας ε, και για την ε, παρουσίαση του πακέτου κυβερνοασφάλειας της Κομισιόν που έχει μεγάλη σημασία για μια λειτουργική ψηφιακή ένωση και έχουμε κάποια συστικό πλαίσιο ακόμα και ζητήματα ποινικού δικαίου. Είναι περίπλοκα θέματα Έχω όμως ένα συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Μιλήσατε για πιστοποίηση. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως είναι το δίκτυο αυτό κέντρων ή κατοτή και Συμφωνώ με την εκτίμησή σας για την ε, ΕΝΙΣΑ. Δεν είναι γνωστή η υπηρεσία και ελπίζω τώρα ότι μέσω της δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Κυβερνοασφάλειας θα μπορέσει και η ΕΝΙΣΑ να έρθει στο προσκήνιο και πρέπει ακριβώς να δείξουμε ότι η Ευρώπη κάνει κάτι στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. Η κυρία Ντελκαστήγιο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μας, την οικονομία μας, την ευημερία μας, η ασφάλεια. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Οπότε, πολύ σημαντική πρωτοβουλία της. Πολύ σημαντικό το ότι αλλάζουν το πρόγραμμα για την ΕΝΙΖΑ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μόνιμη εντολή και χωρίς αναβαθμισμένη συνεργασία. Ομάδα Σίγουρα όλα αυτά βοηθήσουν για την κυβέρνηση ασφάλεια. Βέβαια, το πρόβλημα είναι όλα αυτά να τα καταφέρουμε χωρίς να στερηθούμε ε, ένα ανοιχτό πνεύμα. Υπάρχουν και τέτοιες απόψεις ότι οι αρχέ αυτές έχουν σε σύγκρουση ε, τη δική σας ε, πρόταση. Μπορεί να μα καθησυχάσετε. Ευχαριστούμε κυρία. Κύριε Ζουρίνιο. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, στα πλαίσια αυτού του δομημένου, διαρθρωμένου διαλόγου, θέλω να σας ρωτήσω για την διαδικασία εφαρμογής του Wi-Fi for You. Τι πρόγραμμα επικοινωνίας υπάρχει. Έχετε κάποια στρατηγική για αύξηση συνδέσεων. Έτσι λέει ο κόσμος ότι θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση με κάποια δίκτυα που δεν καλύπτονται. Και όλο ένα και περισσότερη σημασία θα αποκτήσει το πρόγραμμα. δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά για να αναβαθμίσετε την κυβερνοσφάλεια, αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να επιβαλούν κάποιους περιορισμούς στην ελευθερία στο διαδίκτυο. Ήθελα να σα ρωτήσω για το όριμά σα για, για τις παγκοσμίες συμμαχίες. Πρέπει να έχουμε παγκοσμίες συμμαχίε για να διατηρήσουμε το όρεμά μας για την ελευθερία στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε συνάδελφε, λέει ο Ευχαριστώ πρόεδρε και κύριε Κον. Αλλά τι γίνεται και με τα fake news. Η βουλγαρική προεδρεύμα ε, στην άμβλωση και λοιπά, τι βλέπουμε, βλέπουμε διάφορα αρνητικά, όλο αρνητικά, όλο αρνητικά άρθρα τα οποία στριμώχουν ακόμα περισσότερο τις γυναίκες και η κυρία Γιώργα, ε, fake news, αναλυθών ειδήσεων τέλο πάντων στο ίντερνετ. Μπορείτε κάτι να κάνετε και πώς. Ευχαριστούμε συνάδελφε, λέει ο πρόεδρος. Βυρκούνεν. Υπομένει ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωση ανέδειξε τον ρόλο των δεξιοτήτων. Πεςτε μας δύο λόγια παραπάνω, αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Πώς να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Ποιος εν επιγνώση των ε, κινδύνων. Μα κάνει κάτι η Ένωση, μόνο τα κρατημέλη μπορούν να αναλάβουν ενέργειες. Τι είναι με τις ΜΜΕ, γιατί ξέρουμε για τις μεγάλες ε, εταιρείε έχουν ε, πολλούς πόρους, μπορούν να θωρακιστούν για την κυβέρνηση. Έχετε κάποια σχέδια ε, ως Επιτροπή για να βοηθήσετε τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις ε, που είναι πολύ ορθές. Φυσικά αυτή η πρόταση δεν θα φέρει μια θαυματουργή λύση, αλλά εδώ έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς κάποιες κατευθύνσεις. Και θα αντιδράσω επί των συγκεκριμένων ερωτήσεων. Θέλω να επανέλθω στον οργανισμό ΕΝΙΣΑ. Καταρχήν, ε, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα, καθιστώντα ε, μόνο με την εντολή του οργανισμού. Ήταν ε, ο μόνος οργανισμός με προσωρινή εντολή. Πώς θα πείσουμε τους διεθνεί μα εταίρου ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί προτεραιότητα και μακροπρόθεσμη, αν αυτό ο οργανισμός είχε προσωρινή εντολή. Έχουμε επίσης διπλασιάσει τον προπλογισμό και του ανθρώπινου πόρου. Κάθε πρόταση που θα υποστηρίξει αυτή την εντολή είναι ευπρόσδεκτη. Και ήμουν πολύ ευαίσθητη σε σχέση με το θέμα των καταναλωτών. Ναι, ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε με το σύστημα πιστοποίησης. Θα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ε, σε ποιο επίπεδο ασφάλειας ε, ανταποκρίνονται τα προϊόντα τους. Επίσης, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στη βιομηχανία με ένα πιστοποιητικό που θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, όχι μόνο για ένα, σε ένα κράτος μέλος. Είχαμε, ε, χάρη, από τα 150.000 φτάνουμε στα 300.000 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προ τα μπρο. Τώρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να λέμε. Στην πρόταση αυτή δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συνεργασία, όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά και με τη βιομηχανία. Γι' αυτό πριν αποφασίσουμε κάθε ε, πρόγραμμα πιστοποίησης, εμπλέκουμε όλους τους ενδιαφερόμενους. Φυσικά συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να είναι κάποια κράτη-μέλη που θα έχουν το μονοπόλιο. Το ίδιο ισχύει και να μην είναι κάποιες βιομηχανίες που θα έχουν το μονοπόλιο. Γι' αυτό θέλουμε μια δημόσια διαδικασία έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος να μπορεί να συμμετάσχει και μέσω και της Επιτροπής. Πρόκειται για μια πρόταση ιδιαίτερα ευέλικτη λοιπόν. Επιμένω και πάλι στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που θα επιτρέψει να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα συστήματα δίνουμε τη δυνατότητα αυτά που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο να αναπτυχθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, ε, Επίσης ε, έχουμε και το θέμα του νέφους. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την ΕΡΙΝΙΣΑ, να ενθαρρύνει τις ικανότητες των κρατών μελών. Για πρώτη φορά θα μπορεί να το κάνει γιατί θα έχει τις δυνατότητες, τις ικανότητες να βοηθήσει τους λιγότερο αναπτυγμένους. για τον ε, κύριο Κουρουμπάσεβ, για την ερώτησή σας ε, για το θέμα της ενίσα ως οργανισμού. Με ρωτήσατε ότι ε, κάθε φορά που έχουμε μία κυβερνοεπίθεση, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μία αναφορά στον Επίτροπο. Αλλά τώρα εδώ η ΕΝΗΣΑ έχει ένα διαφορετικό ρόλο να διαδραματίσει. Γι' αυτό έχουμε εντός του πεδίου εφαρμογή την ενίσα θέλουμε να έχει μόνιμη εντολή και να επιτελεί επιχειρησιακές λειτουργίες. Δεν μην είναι ένα κέντρο κατάρτισης απλώς, αλλά να μπορεί να αναλάβει δράση και να συνεισφέρει περισσότερο. Έτσι η ΕΝΗΣΑ θα δραματίσει μεγαλύτερο ρόλο και στην πιστοποίηση, στο αποτύπωμα μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό συντονισμό σε περίπτωση επίθεση. Η θα διαδραματίσει ένα ρόλο σε ένα εγχείρημα για την κυβερνοευρώπη. Εμείς θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει κάποιες διαφορετικές ικανότητες, να βρει ποια είναι τα τροτά σημεία των κρατών μελών και να τα βοηθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσουν. Μία άλλη σημαντική πτυχή στη λειτουργία της ΕΝΗΣΑ είναι το εξή. Έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Απάντησης σε περίπτωση κρίσεων. Τώρα προτείνουμε να έχουμε ένα τμήμα εντός ε, του οργανισμού ΕΝΗΣΑ που θα έχει έδρα στις Βρυξέλλες και θα επιτρέπει ταχεία συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών επιχειρήσεων αν χρειαστεί. Αυτή είναι μια πτυχή η οποία μας επιτρέπει να μην αφήνουμε τα πάντα στα χέρια των κρατών μελών μόνο ή μόνο στα χέρια της ΕΝΙΣΑ. Τώρα, για το θέμα της συνεργασίας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διεθνούς συνεργασίας. Προφανώς πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό στην πιστοποίηση προτείνουμε βάση, να βασιστούμε στα διεθνή πρότυπα, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω ένα μοντέλο το οποίο να μπορεί να ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε καλύτερα με τους διεθνείς εταίρους μας. Είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά το αναφέρω σε κάθε διεθνές φόρουμ. Όμω, για να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας ε, για το πόσο σημαντικό είναι πρέπει να κάνουμε και τη δική μας δουλειά, να ενισχύσουμε την εντολή του οργανισμού, να έχουμε ένα σύστημα πιστοποίησης και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αποτελεί μακροπρόθεσμη προτεραιότητα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα του κέντρου αρμοδιοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε όχι μόνο στη τεχνολογία αλλά και στην εμπειρογνωμοσύνη. Υπάρχουν οι εμπειρογνώμονε όμως δεν εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω λοιπόν αυτού του κέντρου ε, ικανοτήτων ε, μέσω και τη δημιουργία και ενό τέτοιου κέντρου εδώ στι Βρυξέλλε. Θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη και να μπορέσουμε να έχουμε ηγετική θέση στο θέμα τη της Ε, Έχω και ένα καλό νέο, κυρία Κάπελ. Ε, θα ανακοινώσω το πιλωτικό πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα στα πλαίσια του 2020, 50 εκατομμύρια ευρώ για να λειτουργήσει ακριβώ αυτό το κέντρο. Και είναι ένα προσωπικό σχόλιο. Δεν θέλουμε ουσιαστικά να μετατρέψουμε τους ανθρώπους ε, σε ε, διαχειριστές της χρηματοδότησης, αλλά θα ήθελα να τους δώσω κίνητρα, γιατί δεν είμαστε εδώ μόνο για να λειτουργούμε κατόπιν των γεγονότων, αλλά να μπορούμε και να αξιοποιήσουμε και την δυναμική που έχουμε για την πρόληψη. σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ε, γνωρίζετε ότι και ως μέλος του Κοινοβουλίου είχα αγωνιστεί για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Όμως, θέλω να αναφερθώ Υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν ε, τεχνικά ζητήματα της κυβερνοασφάλειας και από την άλλη είναι τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει και το νομικό περιεχόμενο. Αυτά φυσικά είναι τρία θέματα τα οποία θα πρέπει να τα παρακολουθούμε σε συνέργεια. Και ε, συνεργαζόμαστε με την Επίτροπο Γιούροβα και με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και τον Αντιπρόεδρο Άνσιπ για τα θέματα αυτά. Ήμασταν ξεκάθαροι για το θέμα του legal contact, ε, για την ε, τρομοκρατική προπαγάνδα, τη ρητορική του μίσους. Ε, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Γι' αυτό το Σεπτέμβριο δημοσίευσαμε μία ανακοίνωση που λέει ότι σήμερα θέλουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην αφαίρεση αυτών των εγγράφων. Το 49% του παράνομου ε, περιεχομένου ε, που έχει εντοπιστεί, συνεχίζει να βρίσκεται εκεί για πάνω από 24 ώρες. Εμείς όμως θέλουμε να δρούμε αμέσως μετά τη δημοσίευση στις 9 Ιανουαρίου συναντήθηκαν διάφορες πλατφόρμες για να... και τους είπαμε ότι θέλουμε περισσότερα αποτελέσματα. Διαφορετικά ε, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε μια νομική πρόταση, μια νομοθετική πρόταση. Για τα fake news ξέρετε ότι έχω δεσμευτεί για το θέμα μετά από σκληρή εργασία τον Νοέμβριο στις 13 Νοεμβρίου ανακοίνωσα